Καλώ ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κοινή συνεδρίαση των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργία περιβάλλοντο. και βιομηχανία έρευνα και ενέργεια. Ξεκινάμε λοιπόν έχουμε τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και ως πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας θα προεδρεύσω στη σημερινή συνεδρίασή μας. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη και αυτό επειδή ο κύριος Λαβία εξακολουθεί να προσπαθεί να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λόγω καθυστέρησης δεν κατάφερε να φτάσει καθυστέρησε η πτήση του. Η κατάσταση είναι παρόμοια με τον κύριο Μπούζεκ. Ο κύριος Μπούζεκ ανέφερε ότι μπορεί ίσως να φτάσει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας και ίσως μπορέσει να προσέθει έγκαιρα στη συνεδρίαση αυτή. Θέλω να σας καλωσορίσω λοιπόν όλους σας. Θέλω να καλωσορίσω τα μέλη των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών που συμμετέχουν και όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχουμε για απόψε, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα. Θα συζητήσουμε για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δάση. Προσήλθε σήμερα και ο Επίτροπος κ. Χόγκαν. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε ότι παρίσταστε και είσαστε εδώ ανάμεσά μας. Και έτσι και η κυρία Κρίστιγκερ είναι επίσης παρούσα ως εισηγήτρια, παρούσα και εκείνη. Πολύ σημαντικό το θέμα, όπως γνωρίζετε, και ίσως θα θυμόσαστε τον Απρίλιο το Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε ένα ψήφισμα για μια νέα πολιτική για τα δάση και για τον δασοκομικό δασοπονικό τομέα συνολικά και είχαμε και μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία που κάλυπτε ακριβώς αυτό το ίδιο θέμα και, και η κυρία Ελίζαμπετ Κέστινγκερ είναι η συγγήτριά μας. Εκτιμούμε πράγματι το ότι είσαστε παρούσα κυρία Κέστινγκερ και η Επιτροπή NVK γνωμοδότησαν για αυτή την έκθεση της κυρίας Κέστινγκερ συνέταξαν γνωμοδοτήσεις και το Συμβούλιο σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε αντίστοιχες ε, παρεμβάσεις όπου η στρατηγική σε σχέση με τα δάση αναφέρεται πρόκειται ουσιαστικά για την αηφόρο διαχείριση των δασών όσον αφορά και το περιβάλλον αλλά και τα κοινωνικά θέματα την κοινωνική πτυχή. Επίσης ε, θα επικεντρωθούμε σε μια καλύτερη επικοινωνία και ε, επαφή όταν πρόκειται για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και της εφαρμογής τους. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε επίσης και ένα πρόγραμμα δράσης ε, για αυτό το τομέα. Ο κύριος Επίτροπος ίσως πιθανότατα θα το αναφέρει αυτό το πρόγραμμα δράσης από πλευρά του. Έχουμε και έναν οδικό χάρτη για την ε, δασική στρατηγική επίσης. Ε, υπάρχουν πολλές προτεραιότητες που έχουν τεθεί και οι πιο σημαντικοί πυλώνες επίσης σε σχέση με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, τούτων λεχθέντων πρέπει να πω ότι έχουμε συμφωνήσει και έχουμε καταλήξει στο να συναντηθούμε απόψε σήμερα. Έχουμε τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές, διότι αφορά αυτό το θέμα και τις τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έχουμε πολλά περιβαλλοντικά θέματα, κλιματικές αλλαγές, έχουμε και την Επιτροπή Βιομηχανίας που εμπλέκεται και εκείνη τα μάλα. Τα δάση είναι μια πολύ σημαντική πηγή βιομάζας. Πολύ σημαντικό αυτό υπό το πρίσμα των βιομηχανιών και των σύναφων δραστηριοτήτων. Σε αυτή την κοινή λοιπόν συνεδρίαση των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αηφορό ανάπτυξη. Επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Γνωρίζω σε σχέση με αυτά τα θέματα το ότι και αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι εδώ σε σχέση με τον κύριο Λαβία και την ε, ε, εκπροσώπηση του. Δεν έχει ζητήσει κάποιο τον λόγο. Ο κύριος Επίτροπος λοιπόν θα λάβει τον λόγο. Κύριε Χόγκαν, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή την συνάντηση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα τάση και τις δασικές εκτάσεις. Ο Επίτροπος ε, Περιβάλλοντος ε, και ε, Επίτροπος Ανάπτυξης είναι επίσης συναρμόδιοι για την στρατηγική αυτή που έχει ως στόχο την βιώσιμη διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία αυτή απαιτεί να συνδυάσουμε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους. Χρειαζόμαστε βιοπικιλότητα, τα δάση μας χρειάζονται επίσης για την παραγωγικότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, αναγέννησή τους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις πολλές αποστολές τους. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δάση είναι σημαντικά για πολλές άλλες πολιτικές, μεταξύ αυτών αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα. Όπως γνωρίζετε τον Σεπτέμβριο ο κ. Γιούνκερ παρουσίασε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 και έθεσε τις 10 προτεραιότητες της Κομισιόν. Και η πρώτη προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις, αύξηση των θέσεων εργασία και ανάπτυξη. Ε, αλλά ε, το περιβάλλον είναι η τρίτη προτεραιότητα ε, πολύ ψηλά δηλαδή και αυτά τα δύο έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζονται στην ε, δασική μας πολιτική. Ε, το κόστος ενέργειας, η, το, η καινοτομία, οι καινούριες δεξιότητες, η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά αποτελούν τμήμα της πολιτικής ατζέντα. Ε, η επικορικότητα και η αναλογικότητα είναι επίση πολύ σημαντικέ. Ε, πρέπει οι δράσει μας να στηρίξουν την βιώσιμη διαχείριση των δασών ε, με συντονισμό των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπου είναι απαραίτητο. Η στρατηγική αυτή αποτελεί μια σφαιρική προσέγγιση όλων των πτυχών που έχουν σχέση με τα δάση και καλύπτεται όλη η αλυσίδα σχετική με τα δασικά προτάσεις και τα δασικά προϊόντα, έτσι ώστε να βοηθήσει ο δασικός τομέας να δημιουργηθούν θέσεις εργασία και να βοηθήσει επίσης και την Ήπεθρο. Ε, η αλυσίδα ε, αξίας ε, σχετική με τα δάση έχει άμεση σχέση με, τα, με τη βιοοικονομία. Ε, θα πρέπει με την καινοτομία να παράγουμε καινούρια προϊόντα και καινούρια υλικά για τον βιοχημικό και άλλους κλάδους. Η βιοοικονομία που βασίζεται στα δάση μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων εργασία. Η βιοοικονομία είναι επίσης ε, πρωτο, ένα ε, ε, από τους πέντε άξονες της κυκλικής οικονομίας. Η καλή είναι ότι ότι τα τελευταία 60 χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός ε, των, του, του, ε, ε ξυλοαποθέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Η, η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στη δράση μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την διατήρηση βιοποικιλότητας και των δασών. Η η πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η βιωσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στην οικονομία μας. Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας ε, συνοδεύεται και πρέπει να συνοδεύεται από την διατήρηση των δασών. Από αυτή την έννοια ε, η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών είναι κλειδί για, ε, για τα βιώσιμα δάση στο μέλλον. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το πλαίσιο συνεργασία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βελτιωθούν και να ανταμυφθούν οι προσπάθειες διατήρησης των οικοσυστημάτων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους διαχειριστές των δασών, με τους ιδιοκτήτες των δασών και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και βέβαια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια ε, έχει ευθύνε και εκτό τη επικράτειά τη. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι προσιλωμένη στην προώθηση τη ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, την καταπολέμηση του υποβάθμιση των δασών και τη απερίμωση, τη αποδάσωση. Ε, ιδιαίτερα δε κατόπιν ε, τη υιοθέτηση ατζέντα ε, του 2030 και τη συμφωνία του Παρισιού. Τα δάση εκεί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μετριασμό τη κλιματική αλλαγή και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι ο, η, η πολυσχηδής, ε, ο χαρακτήρας ε, των, τσιατής των δασών ε, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς μας δράσης. Η διατήρηση των δασών έχει κλιματικά και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη. Επίσης θα ε, η βιωσιμότητα του τομέα μας ε, είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τα ωφέλη των δασών προς την κοινωνία αλλά και να διατηρήσουμε την δυνατότητα να δίνουν τα δάση δουλειά. Τώρα, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Στρατηγική θα ήθελα να σας παρουσιάσω ορισμένο ορόσημα Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και του ενδιαφέρονου φορεί, ανέπτυξε ένα πολιετέ πρόγραμμα ε, εφαρμογή τη ε, ε, στρατηγική με συγκεκριμένε δράσει για την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχου. Οι ενδιαφέρομενοι φορεί επίση συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία εφαρμογή. Τα μέτρα σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξη Πέθρου έχουν ε, αρχίσει να εφαρμόζονται με 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ να προγραμματίζονται ως κρατικές ε, δημόσιες δαπάνες την περίοδο 2014-2020. 2,2 δισεκατομμύρια σε αναδάσωση και δημιουργία δασών. Πάνω από 500.000 εκτάρια θα αναδασωθούν ή θα δασωθούν έτσι ώστε να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή. Πάνω από 200.000 είναι οι δικαιούχοι ε, κατάρτισης, ε, δοκιμών και υπηρεσιών σχετικών με τα δάση. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στην ε, ανεκ, των δασών. Επίσης θα επενδύσουμε στην 800 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην τεχνολογία και σε επεξεργασία, κινητοποίηση, διακίνηση και εμπορία προεδρασικών προϊόντων πριν το τέλος του χρόνου θα ξαναδούμε τα μέτρα, θα τα αναθεωρήσουμε ε, και θα ε, πάρουμε τις νόμες ε, των ενδιαφερομένων στο πλήσιο μιας δημοσίας διαβούλευσης. Ο Horizon 2020 και η εταιρική σχέση για την Ευρωπαϊκή Ενοτομία επίσης δίνουν οικονομική στήριξη στο μέλλον τομέα. Φέτος έχουμε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δάση. Έχουμε ένα focus group για τη διατήρηση βιομάζας, ε, ένα άλλο focus ε, book για τη, ε, faction group για τις νέες αλυσίδες δασικών προϊόντων κλπ που βοηθούν στην υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων. Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, δασικές πρώτες ύλες επίσης θα στηριχθεί. Η Κομισιόν έχει επίση αναλάβει τι εξή ε, δράσει για, τα, για την ξύλια. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια, την, ε, έχουμε στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 ε, έχουμε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη βιώσιμη διακίνηση ξυλίας, για τη χρήση θα ε, εκδώσουμε κατευθείαν γραμμέ για την αλυσιδωτή χρήση της ξυλίας ε, και επίσης ε, σκέφτεται ένα, ένα πρόγραμμα, προγραμματίζει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών. η ατζέντα κοινοτομία επίσης χρησιμεύει. Έχουμε δημοσιεύσει ένα οδηγό για το, ε, περιοχές ε, Natura 2000 ε, όπου προσπαθούμε να φέρουμε σε συνεργασία όλους τους ενδιαφέρομενους φορείς προκειμένου να προωθηθούν συστήματα διαχείρισης και πρακτικές που θα διατηρήσουν τα οικοσυστήματά μας και τα είδη τα οποία είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το διεθνή πυλώνα, <clears throat> βρισκόμαστε, είμαστε πρωτοπόροι πόροι στην κάλυψη νομικών κενών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εμπορία ειδών ξυλίας. Ε, η, η έναρξη της FLAG, ε, πρωτοβουλίας FLAG στην Ινδονησία είναι σημαντικό γεγονός. Στηρίζουμε επίσης αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, για την εφαρμογή διεθνών κανόνων προστασίας και διατήρησης των δασών η Κομισιόν, σύμφωνα με το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, ε, σκοπεύει να ε, κλιμακώσει τις προσπάθειές της. Μια μελέτη, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο πρόγραμμα δράσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποδάσωση. Πιστεύω ότι αυτά τα ορόσημα, τα οποία μόλις σας παρουσίασα, αποτελούν σημαντική όθηση για την βιώσιμη διαχείριση των δασών, για τον πολιτορικό χαρακτήρα τους, αλλά και πάλι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Θα ακούσω τη συζήτηση και θα επανέλθω στο τέλος ε, με παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Επίτροπε Χόγκαν για την εισαγωγική σας αυτή παρέμβαση. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία τώρα στα χέρια μας για να κάνουμε μια συζήτηση. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ομιλητών. 1,5 λεπτό θα δώσω στον καθένα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε μέχρι τις 8.30. 1,5 λεπτό λοιπόν έκαστος. Θα βλέπετε και το χρόνο. Κυρία Κιώστιγκερ, η συγγήτριά μας, έχει το λόγο για μισό λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ Επίτροπε που σήμερα έχετε την ευκαιρία, έχουμε την ευκαιρία από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας να συνέλθουμε και να συζητήσουμε είναι πολύ σημαντικά αυτά σε σχέση με τα συνοδευτικά όσα γίνονται στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε εδώ από το Κοινοβούλιο να μπορέσουμε ίσως να ασκήσουμε την επιρροή μας. Για τη στρατηγική αυτή πάντα ήταν σημαντικό για μας πάντα η σωστή προσέγγιση όσον αφορά τα δάση. Υπάρχουν πολλές νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, και έχουμε μέσα στο πλαίσιο όλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, ε, έχουμε την επιρροή που πρέπει να ασκηθεί για την πολιτική και πιστεύω ότι αυτά που εμείς όλοι από κοινού πάντα διαπιστώναμε είναι ότι η δασική πολιτική συνολικά στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Έχουμε χώρες όπως τη Φινλανδία και την Αυστρία. Έχουμε χώρες ε, που στο παρελθόν έκαναν πολλά σφάλματα και τώρα εξαρτώνται από εισαγωγές από τρίτα κράτη για την ξυλία τους και έχουμε άλλα κράτη που έκαναν πολλά, έπραξαν πολλά όσον αφορά προγράμματα και με θετικά αποτελέσματα. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα ισοπεδωτικό μέτρο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί στην πολιτική και υπάρχουν οπισθοδρομήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν η αηφορία να λαμβάνεται υπόψη συνολικά για την δασοκομεία δασοπονία. Έχουμε το Forest Europe ε, με την αηφορία και βιωσιμότητα στην ανάπτυξη, με την πιστοποίηση όσον αφορά την ξυλία. Όλα αυτά πρέπει να συνεχιστούν και είναι σημαντικά ώστε στη στρατηγική για τα δάση να τηρείται, ώστε να λαμβάνετε υπόψη από τα κράτη το θέμα και της πιστοποίησης, αλλά να μην δημιουργούνται πάντα παράλληλες ε, δομές ε, με επικαλύψεις. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε θέματα ανάργειας. Και εδώ το δάσος και η δασοπονία, δασοκομεία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Από την, ε, την αντίστοιχη γενική διεύθυνση πρέπει να υπάρξει επαρκές στελεχειακό δυναμικό ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να λαμβάνουμε υπόψη τις νομοθετικές πρωτοβουλίες όταν αυτές ε, αναφύονται και για την εφαρμογή τους. Και πρέπει αυτό το οποίο ζητήσαμε, μια στρατηγική για τα δάση με αναβάθμιση, αναβάθμιση της Επιτροπής Δασών με τους ε, πραγματογνώμονες εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δούμε δηλαδή πώς αυτά τα αιτήματα υλοποιήθηκαν. Εν τέλει έχουμε και μια δημόσια κρόαση που έχει προαναγγελθεί Σήμερα θα ήθελα να κάνω την πρόταση οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας να μπορέσουν αυτή την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συμμετοχή πραγματογνωμόνων να συμμετάσχουν σε αυτή. Αυτό είναι κάτι το ευκταίο και επιθυμητό διότι υπάρχουν διαφορετικές ενώσεις συμφερόντων που μπορούμε να ακούσουμε τις απόψεις τους και μπορούμε έτσι να τους δώσουμε ένα βήμα για να εκφραστούν. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτής της συνεδρίας απόψε. Ευχαριστώ. Κυρία Μίλερ. Σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε για τα όσα μας αναφέρατε. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ότι τα δάση και η δασοκομεία, δασοπονία συζητώνται όλα από κοινού μεταξύ μας απόψε είναι σημαντικό σε σχέση με τη γεωργία και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πραγματικά ακολουθούν μια αϊφόρο πολιτική και δράση σε σχέση με τα δάση πρέπει πραγματικά να προστατευτούν και αυτοί και οι καταναλωτές. Όπως και η προλαλή σας, έτσι και εγώ λέω ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορε... διαφορές στα κράτη-μέλη, διαφορές στις προσεγγίσεις και στην υλοποίηση όλων αυτών. Από τα κάτω προς τα άνω πρέπει πραγματικά να αναπτυχθούν αυτές οι προτάσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη αηφόρο δασοκομεία στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό από πλευράς του τομέα της ε, ε, πιστοποίησης να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα να μην ε, υπάρξει διασπάθηση πόρων και να μην υπάρξει παρέκκληση από τους στόχους. Απορρίπτουμε λοιπόν μια τέτοια κατακαιρματιστική προσέγγιση. Ένα παράθυμα από ε, τον καθηγητή Ντέρκα ως από το 2007 που ε, αναλύοντας το μέλλον είπε αν υπάρχει ένας ανταγωνισμός ε, για την αηφορία, ποιος ξέρει ποιος θα κέρδιζε στο τέλος. Ελπίζω λοιπόν ότι υπό αυτό το πρίσμα θα καταλήξουμε στην βέλτιστη στρατηγική για τα δάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε Χόγκαν, που ήρθατε για να μιλήσουμε εδώ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ και την κυρία Κέστιγκερ και την κυρία Μιούλερ που μας ε, παρουσίασαν το θέμα και πήραν κάποια από τα λόγια από το στόμα μου. Θα μιλήσω για κάποια άλλα θέματα. Θα πω κατευθείαν στο ψητό, λοιπόν. Θα μιλήσω για την αρχή τη αλυσιδωτή αντίδραση, του cascading. Εμεί, οι νομοθέτε, προσπαθούμε να νομοθετήσουμε το πώ και το γιατί ένα γεωργό ή ένα που ασχολείται με το δάσο θα πουλήσει τα προϊόντα του σε οποιονδήποτε. Εν συνεχεία, πηγαίνουμε στου ιδιοκτήτε γη και λέμε ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο ε, χρήση του δάσου σα. Λε και είναι. Ε, δημόσιο αγαθό. Όμως μην ξεχνάμε εδώ πέρα και την ε, ιδιωτική κατοχή γης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, επίσης μιλάμε για τα δάση, ε, λες και έχουν όλα τα ίδια δέντρα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, η λεγόμενη βιοοικονομία, που αναπτύσσεται ταχαίω στη Φιλανδία, ε, Αυστρία και αλλού. Και εκεί είναι η ποιότητα τη ύνα που μετράει. Ένα δέντρο μπορεί να φτιάξει χαρτί, ε, ρούχα, ε, ενέργεια, καύσιμα, χημικά. Διερωτώ με, Επίτροπε, πώς θα μπορέσετε να κάνετε μια πρόταση η οποία θα λάβει υπόψη τη διαφορετική ποιότητα που μπορεί να έχει η κάθε ίνα του δέντρου. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης ή η αγορά να αποφασίσει σε ποιον θα πουλάει ας πούμε, το προϊόν του και ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης του δάσους αυτού. Ζητώ συγγνώμη που θα σας ξυπνήσω λιγάκι. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι η Κομισιόν δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα δασοκομεία. Δεν το αναφέρει η συνθήκη. Ο Επίτροπος όμως ενθαρρύνθηκε ίσως από την ψήφο στην Ολομέλεια που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες που του λέγαμε με αυτόν τον τρόπο να κάνει κάτι για τα δάση αλλά αυτή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν, είναι, δεν αποτελεί αναθεώρηση των συνθήκων και επομένω. δεν θα έπρεπε να είμαστε καν εδώ να συζητάμε αυτό το θέμα. Ενθαρρύνουμε στην πραγματικότητα τον Επίτροπο να νομοθετεί σε τομεί που δεν έχει αρμοδιότητα. Ζητώ συγγνώμη. Δεν σα αρέσει η αλήθεια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνο τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρηματοδοτήσει τι πρωτοβουλίε για τη δασοκομεία είναι μέσω των προγραμμάτων άπευση υπαίθρου. Αλλά αυτά θα πρέπει να προσδιοριστούν σε επίπεδο κρατών μελών. Και αν το κράτο μέλο δεν καθορίσει μία συγκεκριμένη δασική πρωτοβουλία, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εμπλακεί καθόλου. Μην το ξεχνάτε ότι στην πραγματικότητα προχωρα... πατάτε σε πολύ επικίνδυνα νερά. Επίσης με ανησυχεί ότι με φτρασή τρόπο ο Επίτροπος, ας πούμε, ε, μιλάει για μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης ε, που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, η φύτευση, ας πούμε, ε, δέντρων. Ε, μην ξεχνάμε ότι τελικά αυτά τα δέντρα, αν έχουμε πάρα πολλά από τέτοια δέντρα, ας πούμε, στην πραγματικότητα ή θα... Ναι, με στην αρχή απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά μετά κάποια στιγμή, ας πούμε, καταστρέφονται, σαπίζουν, ας πούμε, και κλείουν ε, διοξείδιο του άνθρακα πίσω στην ατμόσφαιρα. Δεν μπορεί να σταματήσει τη φύση. Ε, ευχαριστώ. Είμαστε πολύ συνηθισμένοι στα καμπανάκια που μας σημαίνεται. Και αυτά τα ψυχρά ντους που μας, ε, με τα οποία μας ρένεται μερικές φορές ε, είναι χρήσιμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, στην κοινή μας αυτή συνεδρίαση. Είναι πολύ σημαντική η συνεδρίαση αυτή. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα περιοριστώ σε ένα θέμα της δασικής ε, στρατηγικής. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των δασών για την ε, δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα στην παγκόσμια πολιτική και στην ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το τομέα. Έχουμε συμφωνίες ε, στο Παρίσι, έχουμε τη συμφωνία στο Μαρακές και επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι όλοι θέλουν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να χρησιμοποιήσουμε τα δάση, ούτως ώστε λοιπόν να περιορίσουμε τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα. Όμως, σε ό,τι αφορά την κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τάση μας είναι πολύ πιο... και η προσπάθειά μας είναι πολύ πιο απαιτητική και αυστηρή από την προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η δική μας προσέγγιση είναι κατά τη διαφορετική. Ίσως οι κανόνες που προσπαθούμε να αναπτύξουμε τώρα θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βοηθήσουμε αυτές τις δύο προσεγγίσεις ώστε να συγκλίνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντιφάσεις. Ε, ο Επίτροπος είδε τις διαφορές μας. Υπάρχουν δύο α, τάσεις εδώ. Ο Στιούαρτ ε, εξέφρασε τη μία. Ε, το μόνο ακριβές που είπε είναι αυτό για το καμπανάκι. Η δασοκομεία δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κλιματική αλλαγή είναι και αυτά τα δύο πράγματα κάπου εφάπτονται. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητα. Ε, τελικά το ένα είναι πιο σημαντικό από τα άλλα. Και νομίζω ότι η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι πολύ πιο σημαντικό από τα δάση. Τα δάση μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς και γενικά η χρήση των, της γης, ας πούμε. Ε, και σας ενθαρρύνω να ασχολείστε με την δασοκομεία και με όλα τα θέματα που αφορούν την δασοκομεία και με όλα τα θέματα εξάλλου που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Προσοχή, προσοχή λοιπόν εδώ. Δεν το ε, συνειδητοποίησα μέχρι να διαβάσω όλο το κείμενο. Όλοι είμαστε υπέρ ενός ε, υπέρ της φύτευσης περισσότερων δασών για πολλούς λόγους, αλλά παραδείγματο χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, υπάρχουν περισσότερα, περισσότερο αποθηκευμένο διοξίδιο του άνθρακα στα δενδρύλια, ας πούμε, από ότι στα δάση πολλών άλλων χωρών. Επομένως, προσοχή, προσοχή. Ε, να μην τα μπερδεύουμε όλα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ε, πράγματι δεν έχουμε πολλές αρμοδιότητες σε δασικά θέματα, δυστυχώς. Όμως ε, έχουμε λύσεις για να καλύψουμε τα κενά της έλλειψης ε, δασικής πολιτικής στην Ευρώπη. Το να ενισχύσουμε μια σφαιρική προσέγγιση όπως το προτείνει η Κομισιόν με την οικονομική και δασική διάσταση είναι σωστό. Τα δάση δίνουν δουλειά στους ανθρώπους υπαίθρου. Δεν είναι απλώς όμορφα ε, ή απορροφούν απλώς διοξείδιο του άνθρακα. Δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Ε, δεν μπορούμε όμως να χρηματοδοτούμε τη δασική πολιτική μέσω του Ταμείου ε, Ανάπτυξη Πέθρου. Εκεί τα ποσά είναι μικρά, θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης. Ε, λίγοι πόροι, λίγα τα κονδύλια, αλλά επιπλέον τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ε, πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξη Πέθρου. Ε, στην πραγματικότητα θα χρειαζόμαστε με πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική δασών. Πάντοτε ε, η χρηματοδότηση ήταν ανεπαρκής. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε οι αγρότες να συνεχίσουν να ζουν στην ε, Ήπεθρο, να μην εγκαταλείπουν τις ε, γέες τους και να αποφύγουμε την αποδάσωση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ακολουθείτε τη σωστή άγουσα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, κύριε Επίτροπε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας, Επίτροπε. Πράγματι, στο Παρίσι και στο Μαρακές πολλοί άνθρωποι κάνουν λόγο για τον ρόλο των δασών και της κλιματικής πολιτικής και έχουμε και προτάσεις όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών ρήπων, όσον αφορά τους βιομηχανικούς τομείς. Γι' αυτό τα δάση θα διαδραματίζουν σίγουρα ένα σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, αυτό είναι ακόμα συμβολικό, συμβολικού χαρακτήρα μέχρι, μέχρι σήμερα. Το ποσοστό απορρόφησης μπορεί να μετράται και ως ποσοστό ή τμήμα εθνικής πολιτικής μείωσης εκπομπών των ρήπων αλλά επίσης και ως τμήμα της δασοκομικής πολιτικής. Αυτά όμως δεν είναι ικανοποιητικά ως λύσεις για χώρες που έχουν μεγάλα δάση. Μια τέτοια χώρα είναι η Πολωνία. Και εδώ σε σχέση με τον ρόλο των δασών που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ενεργειακό μείγμα, αυτό θα τροποποιούσε τους δείκτες για την ενεργειακή πολιτική στη χώρα μας. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα έπρεπε να αυξηθούν τα κατόφλια, τα επίπεδα σε σχέση με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη Συμφωνία Παρισίων και συμφωνείτε με τον Επίτροπο Κανιέτε ότι είναι το μέγιστο αυτό το οποίο μπορούσε να συμφωνηθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Πέτης έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δείχνετε ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ επίσης ε, για την επαφή και συζητήσεις που διεξάγεται μαζί μας ε, απόψε που είναι η τρίτη φορά νομίζω για αυτό το σημαντικό θέμα. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα, τη δασοπονία και κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους, τους φυσικούς τους πόρους με υπεύθυνο τρόπο. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για την ενέργεια, για την οικονομία και βρίσκεται καθοδόν και ε, μια δέσμη μέτρων για την ε, αηφορία στην ε, δασοκομεία. Όλα τα κράτη πρέπει να δούμε την θέση στην οποία βρίσκονται και πρέπει να δράσουν ε, με ενιαίο τρόπο, άσχετα αν έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό δασικής κάλυψης. Θα πρέπει να ληφθούν ε, αυτές οι ιδιομορφίες και διαφορές υπόψη. Διαφορετικά χώρες που έχουν ένα δυναμικό δεν θα τύχουν ε, αρκετό κινήτρο. Η Κροατία έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης δασών όπως και άλλες χώρες ε, ε, προς τον, ε, στην κοιλάδα του Δούναβη. Έχουμε λοιπόν το δυναμικό αν όλα τα κράτη-μέλη βρεθούν στο ίδιο επίπεδο λοιπόν και από το ίδιο επίπεδο εκινήσουν η αηφορία στη διαχείριση των δασών δεν θα λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Όλα τα, τα δέντρα που ξυλεύονται που υλοτομούνται θα πρέπει να μας κάνουν να εξετάσουμε την αηφορία ακριβώς ε, στα δασοκομικά. Διαρωτώ με πώς σκοπεύετε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χέσλινγκ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τη δυνατότητα διεξαγωγή αυτή τη συζήτηση. Είναι θετικό να μπορέσει να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά κάποιε πτυχέ βλέπω ότι δεν καλύπτονται επαρκώ. Τα δάση πλήττονται από τις κλιματικές αλλαγές τα μάλιστα και χρειαζόμαστε προσαρμογές και τροποποιήσεις για την αηφορία, για τη διατήρηση των ε, δασών. Δεν υπάρχει όμως μία και μόνη απάντηση ε, για την Ευρώπη. Είναι πολύ διαφορετική εικόνα των ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει μια προσαρμοσμένη στρατηγική να ακολουθηθεί για να πετύχουμε την ε, αηφόρο διαχείριση και πρέπει εδώ και το θέμα της βιωσιμότητας όχι μόνο για την ξυλία να εξεταστεί, αλλά και για την πολιτική βιοπικιλότητα και ποικιλομορφία. Πρέπει να συνεισφέρουμε λαμβάνοντα υπόψη τη συνεισφορά του δάσου και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στην ξύλευση, στην υλοτομία. Επίση, και η χρήση και η μεταποίηση, ε, εκμετάλλευση των ε, δέντρων. Πρέπει εδώ να δούμε, δεν είναι δυνατόν να καίγονται μόνο τα δέντρα, είναι η πιο θα έλεγα ε, η λιγότερο αηφόρος ε, εκμετάλλευση, είναι μια χαζή εκμετάλλευση. Πρέπει εδώ να δούμε συστήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στην Ευρώπη για να υπάρξει αηφορία. Εδώ σε σχέση με τα δάση πρέπει να συνεισφέρει η Ευρώπη για την αηφορία τους. Μία τελευταία παρατήρηση επίτροπε και πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο και σε χώρες εκτός Ευρώπης ε, γίνεται όσον αφορά την εκμετάλλευση των δασών. Για παράδειγμα, σε σχέση για παράδειγμα και την καταστροφή δασών που ακολουθείται από κάποιες χώρες για την παραγωγή τροφίμων, την καλλιέργεια δηλαδή σε αρρώσιμες γέες ε, για να υπάρξει παραγωγή τροφίμων. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία τη κοινή συνεδρίαση των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών παρουσία του κ. Χόγκαν, γιατί το θέμα είναι οριζόντιο, αφορά την οικονομία, το, το περιβάλλον και τα θέματα τη υπαίθρου. Πολύ σημαντικά. Το δάσο, το ξύλο δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, δεν το προβλέπει η συνθήκη και δεν αναφέρεται στη γεωργική παραγωγή. Επομένω είναι κρατική αρμοδιότητα. Όμως νομίζω ότι είναι χρήσιμο, για να πω απαραίτητο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγύψει επί του θέματο αυτού, γιατί το θέμα της ανανέωσης μπαίνει εδώ και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι για να διευκολύνει την ανανέωση. Όχι μόνο στο, στα εδάφη των κρατών μελών τη ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα πλαίσια τη συνεργασία που έχει, ειδικά με την Αφρική και μην ξεχνάτε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα μπορούσε να προωθήσει τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Μπορούμε να σκεφτούμε ε, την επανεμφύτευση. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να το ξεχάσουμε και να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης, κύριε Επίτροπε. Το ξύλο είναι φυσική ύλη, ζωντανή ύλη. Ε, μπορεί να δώσει όμως πλοία πάρα πολλά νέα προϊόντα με τελείως διαφορετική χρήση. Αυτά τα δύο σημεία λοιπόν θα πρέπει να τα κρατήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παρούσα στην ε, διαχείριση των δασών στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις για τον Επίτροπο που έχουν να κάνουν με την αποψήλωση των αναπτυσσόμενων λεγόμενων χωρών γιατί και επίσης για το φινικέλαιο που σχολίασε ο συνάδελφος. Ξέρετε ότι χρησιμοποιείται αυτό το λάδι σε μεταποιημένα προϊόντα, σε, σε γεωργοκάψιμα, ε, ο, οδηγεί στην Ινδονησία, στη Μαλαισία και σε άλλες χώρες σε φο, φοβερή αποψήλωση. Ε, τι άποψη έχετε κύριε πίτροπε. Αυτή η καταστροφή του συστήματος των πιστοποιητικών για το φινικέλιο. ε, τι γνώμη έχετε για αυτήν, ε, πώς μπορείτε να σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο και στο επίπεδο Παρισιού, και στο IG. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τις δηλώσεις που κάνετε πριν λίγο. Για το κρέας, είχατε πει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την κατανάλωση και παραγωγή κρέατος. Ε, είπατε ότι θα βάλετε 15 εκατομμύρια ευρώ για να προωθήσετε αυτή την ε, κατανάλωση κρέατος. Η, παραγωγή κρέατος στη Βρασιλία, ας πούμε, ε, οδήγησε σε αποψήλωση δασών. Ε, αυτή τη στιγμή η κατανάλωση κρέατος προκαλεί το 15 με 20% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας ε, που αναλάβετε στο Παρίσι. Πώς μπορείτε να είστε συνεπείς. Από τη μία έχετε τη λεγόμενη βιώσιμη στρατηγική για τα δάση και από την άλλη έχετε αυτές τις δηλώσεις. Πώς γίνονται αυτά, πώς πάνε μαζί. Ο κύριος Άντριου, ε, ευχαριστώ Επίτροπε που παρουσιάσατε την δασική στρατηγική στις τρεις επιτροπές. Πολλά στοιχεία ακούστηκαν ήδη. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι για το θέμα των αρμοδιοτήτων και τα όρια της δασικής στρατηγικής της Κομισιόν, δεδομένων των ευθυνών που έχει το κάθε κρατός μέλος. Το να λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία δασική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο δασικός πλούτος ε, είναι διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να μιλάμε για δασικές στρατηγικές ε, είναι ένα κοινό υπόβαθρο το οποίο έχει να κάνει με το κλίμα και την προσπάθεια που κάνουμε για το κλίμα. Ε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δάση στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο με την Νότια Ευρώπη, με τα δάση στη Νότια Ευρώπη. Πολλέ ερωτήσει ακούστηκαν βεβαίω. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να δούμε ξανά το θέμα της ανάκτησης δασών ε, το θέμα της αγροδασοκομείας που τέθηκε επίσης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα στο μέλλον. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Εσείς, αυτό το πολιετές σχέδιο για την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής, των δασικών στρατηγικών, πώς το προσδιορίσετε, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητας της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης και πώς το δάσος θα μπορούσε να είναι ε, μοχλός τοπικής ανάπτυξης να οδηγήσει σε τοπική ανάπτυξη. Και στα πλαίσια της κλιματικής, τη άφηση δημοκρασία του πλανήτη, η δασική στρατηγική τι, προβλέπει, τι προβλέπει πολύ συγκεκριμένα, ούτω ώστε να συνεισφέρει πολύ συγκεκριμένα στην ανάσχεση της αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε συμφωνούμε με την ανάπτυξη σε σχέση με την αηφορία. Είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της βιοπικιλότητας ε, για να διατηρηθεί ε, η δασοπονία και θα ήθελα επιπλέον να πω ότι σε σχέση με τις ε, ε, αρρώσιμες γιές, τις ε, καλλιεργήσιμες γιές, πρέπει να αποφύγουμε την μονοκαλλιέργεια και όπως συμβαίνει στην Γαλλικία ή όπως συμβαίνει και στην Πορτογαλία, για παράδειγμα με τους ευκαλύπτους και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μαζικά λιπάσματα και ε, αγροτοξικές ουσίες. Πρέπει να μπορέσουν να γίνουν σεβαστές ε, οι αρχές της αηφορίας ε, όσον αφορά αυτού του είδους τις εκτάσεις και καλλιέργειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θέλω για άλλη μια φορά να επανέλθω στο θέμα της βιομάζας από ξυλία Υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά την, την Ευρώπη. Πολλά μικρά προγράμματα υπάρχουν όπου χρησιμοποιείται βιομάζα με αυτά για θέρμανση εγώ ως δήμαρχος όταν ήμουν δήμαρχος ε, ένα, μια μονάδα καύσης ε, ε, είχαμε δημιουργήσει με την ξυλία που χρησιμοποιούσαμε μέσω καύσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα θέρμανσης. Θέλω να ακούσω κόδωνα κινδύνου να μην ανοίξει τώρα η δυνατότητα πιστοποίησης που τίποτα άλλο δεν θα κάνει που θα δημιουργήσει εταιρείε πιστοποίησης που θα βγάζουν τα λεφτά τους εις βάρος ε, εκείνων που δημιούργησαν ε, σε μικρότερη κλίμακα ε, κάποιοι επιχειρηματίες. Εξάλλου πρέπει να δούμε ότι είναι πολύ, μικρής κλίμακας τέτοιου είδους μονάδες. Για τη νέα πιστοποίηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επανέλθω σε όλα τα ζητήματα τα οποία έθιξαν οι συνάλφοι πέραν της ανάγκης προστασίας των δασών και τη σημασία τους για την βιοπικιλότητα, ε, τον πολιτορικό χαρακτήρα τους, ε, το γεγονός ότι δίνουν θεσσαρασίας, οπότε συνεισφέρουν στην οικονομική δραστηριότητα της υπαίθρου, όλα αυτά τα είπαν οι συνάδελφοι. Επίση τη σημασία τους στην ανάπτυξη πέτρου. Εγώ θα σταθώ σε τρία θέματα. Και αυτό ελέγχθη βέβαια, αλλά θέλω να το επαναλάβω. Η στρατή και τα δάση τις δασικές εκτάσεις θα πρέπει να ενταχθεί ε, μάλλον σε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να ενταχθεί η μεγάλη βιοπικιλότητα της, των ευρωπαϊκών δασών. Ε, η βιοπικιλότητα στην Ευρώπη είναι διαφορετική από τη βιοπικιλότητα σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δείξουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φέρουν αποτελέσματα. Δεν είναι απλώ υποχρεωμένα να ε, διαθέτουν τα μέσα, αλλά να παίρνουν αποτελέσματα. Η κλιματική αλλαγή από την άλλη μεριά επιδράσει όλα τα δάση. Ιδιαιτέρως στους ζώντες οργανισμούς, ε, χλωρίδα και πανίδα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, την κλιματική αλλαγή λοιπόν και την επίδρασή της στα δάση και τους ζώντες οργανισμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, υποβάθμιση του εδάφους. Τέλος, να επιθυμώ η Κομισιόν, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, να σηκώσει τα μανίκια και να πιέσει τα κράτη-μέλη, γιατί οι δασικοί μας πόροι θα πρέπει να προστατεύονται παρόλο ότι, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Κύριε Επίτροπε, σε σχέση με τα δάση υπάρχουν ίσως ε, διαφορές αλλά μπορούμε ίσως κάπου να συμφωνήσουμε με ανησυχεί ότι στη νέα δασοκομική στρατηγική με τα σημεία που ζητείτε να υλοποιηθούν όσον αφορά το υλικό για οικοδομικές εργασίες και για συσκευασίες ζητήσαμε στη επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει τον τομέα αυτό για την συγκεκριμένη χρήση ξυλία ε, σα στον οικοδομικό τομέα. Δύο ερωτήσεις. Στα κράτη-μέλη, μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα στον οικοδομικό τομέα, ε, υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες ε, σε σχέση με την οικοδόμηση με ξυλία. Αν δημιουργήθηκαν τέτοιες δυνατότητες, ποιες είναι αυτές σε σχέση με μια επισκόπηση, εξέταση, έγινε κάτι, κινητοποιήθηκε η αγορά και ο οικοδομικός τομέας με χρήση ξυλίας. Άλλη ερώτηση. Πώς βλέπετε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Επίτροπε, σε σχέση με τις οργανικές ε, ενώσεις ε, και την χρήση αυτών. Πώς το βλέπετε και πώς το αντιμετωπίζετε. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το σκυρόδεμα και τα προϊόντα χαλιβουργία να μπορούν ίσως να χρησιμοποιούνται καλύτερα σε σχέση με αυτού του είδου τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, στο τέλος των όσων μας εκθέσατε, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα δράσης για την Ινδονησία. Είχα, θα είχα μία ερώτηση. Στην Ινδονησία ακολουθείται ισχυρή αποψήλωση, έντονη αποψήλωση δασών και έχουμε και τις ε, φοιτίες ε, φοινικέλεου. Δεν μπορώ να δω πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς είναι δυνατόν με ένα πρόγραμμα δράσης να αναχαιτιστεί αυτή η κατάσταση και με τις κλιματικές αλλογές ε, να δούμε τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ευρώπη. Αναφερθήκατε για μεγάλα ποσά όσον αφορά την προαγωγή κρέατος. Ε, για την παραγωγή αυτού του κρέατος ε, δημιουργούνται όλες φυτίες σόγιας, αποψηλώνονται δάση Πώς μπορούν όλα αυτά να ευθυγραμμιστούν με μια στρατηγική καταδάση που θα είναι αηφόρος όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπόθηκε επανειλημμένως ότι η δασική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως Πολλέ αποφάσεις λαμβάνουν σε ευρωπαϊκό πεδίο και επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές για τα δάση και τι δασικέ εκτάσεις. Και αυτές οι αποφάσεις πολύ συχνά δεν συνάδουν με την ε, στρατηγική μας για τα δάση. Η στρατηγική για τα δάση είναι ισορροπημένη, αλλά υπάρχουν τρεις πρωτοβουλίες που συζητώνται ή θα συζητηθούν σύντομα. Το Λουλουσιεφ, η διοδηγία της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας και, και αυτή για την στρατηγική για τη βιοοικονομία. Μια και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα μιλήσω για την ε, χρήση της ε, γης και την αλλαγή της χρήσης της γης και τα δάση. Το 75% το, του εδάφους μας είναι δάση στη Φιλανδία, από την οποία προέρχομαι. Η Φιλανδία λοιπόν είναι ένα μεγάλο δάσος. Οι πολίτες μας ε, είναι προσιλωμένοι στη μείωση των εκπομπών, αλλά τα δάση είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και για άλλους λόγους, για, για την οικονομία μας και για κοινωνικούς λόγους. Το οποίο σημαίνει ότι επιθυμούμε βιώσιμη δασοκομεία στη Φιλανδία. Τώρα, η Λούλου πρόταση Λούλου Σιεφ για τη χρήση της γης αποδεικνύει ότι ο, ο ρόλος της βιώσιμης διαχείρισης ε, των δασών στην ε, καταβολή δεν είναι σαφής. Ε, ο δασικός τομέας ε, δεν διατηρεί απλώς αυξημένη απορρόφηση ε, διοξείδιο του άνθρακα, αλλά δίνει και δυνατότητα παραγωγής βιοπροϊόντων. Επίσης, ε, μας δίνει καινοτόμους τρόπους για να πολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ε, συνεπώς, η βιώσιμη ε, δασοκομεία έχει τεθεί σε κίνδυνο από την πρόταση Λουλουσιεφ. Αυτό ήθελα να το πω, αυτό ήθελα να πω στον Επίτροπο. Um, thank you very um, Ευχαριστώ. Κίνδυνο τη απομόνωση τη υπαίθρου. Τι έχει να πει ο Επίτροπο γι' αυτό, ιδιαίτερα στην ε, δυτική και βορειοδυτική Ιρλανδία, όπου εξαιτία ε, γεωργικών πρακτικών, των και, ε, μείωση των τιμών κλπ. Ε, ε απεριμώνεται η ύπεθρος και τελικά δεν θα μείνουν άνθρωποι στην Ήπεδρο ή θα είναι μικρές κοινότητες. Σε ό,τι αφορά την τελευταία γνώμη, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας γνώμη για την ε, πρόταση Σιεφ και τη σχέση με τη στρατηγική για τα δάση. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι τα λογιστικά συστήματα, μάλλον τα συστήματα καταγραφής σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την πυκνότητα της ξυλίας. Στην Ιρλανδία έχουμε το εξή πρόβλημα. Ε, πολύ συχνά κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ξυλία δεν είναι αυτή η οποία είχε παραγγελθεί, αυτή που αναφέρεται από τις αρχές ε, και έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη στον κλάδο. Ε, θα μπορούσε να γίνει μια ευρωπαϊκή έρευνα τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια, ε, ένα κομμάτι στρατηγική έτσι ώστε να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη ε, των πολιτών ότι αγοράζουν δηλαδή την ξυλία η οποία αναφέρεται στη συσκευασία. Επίσης για το θέμα των αρμοδιοτήτων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλώ για αυτό το θέμα, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τη ΣΥΤΑ. Ε, ποια είναι η προτεραιότητά μας τελικά. Thank you. This is very good priority Πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα που φέρατε τρει επιτροπέ. Χαίρομαι που ο Επιτροπό ήρθε εδώ μαζί μα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιο έχει αρμοδιότητα, ε, αλλά τον, το ότι συμφωνήσαμε μαζί για την δασική στρατηγική και μιλήσαμε για τον ε, πολυσχηδή ρόλο των δασών μας για την, ε, και για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών που μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Η δασοκομεία όταν λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο είναι πολύ καλύτερη ε, και για το θέμα της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Εγώ είμαι στην Ήτρε και ετοιμάζουμε ένα έγγραφο. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι πολιτικές μας να είναι συνεπείς πολιτικές όπου εμπλεκόνται τα δάση. Ε, η Λουσιέφ είναι πολύ επίκαιρη πολιτική. Υπάρχει και η αναθεώρηση της πολιτικής αλλά και το ενεργειακό πακέτο Θέλω να υπάρχει συνάφεια σε όλε αυτέ τι πολιτικέ. Ε, την Κυριακή Στήλιαν στο μέλλον οι τρει επιτροπές να συνεργαστούν για το θέμα των δασών. Το πακέτο για την ενέργεια επίσης έχει κάποια βιώσιμα κριτήρια. Το ίδιο ξύλο το οποίο ε, υπάρχει ε, στο δάσος ε, φτιάχνει ε, ρούχα, φάρμακα, χαρτί κτλ. Και τα υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενέργεια. Το 40% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προέρχονται από το ξύλο. Δύο σύντομες ερωτήσει. Τα δεδομένα για τα δάση μας στην Ευρώπη δεν είναι αρκετά καλά. Έχετε τίποτα καλά νέα θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα για τα δάση μας. Ε, η βιοοικονομία και η, στρατηγική, η αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιοοικονομία. Μετά από όλες τις προσπάθειες που κάναμε στον ορίζοντα 2020 και στο ΕΦΙΣ, καλό θα ήταν να έχουμε μια νέα στρατηγική ε, για τη βιοοικονομία, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα χρησιμοποιεί πια ορυκτά καύσιμα. Ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε που παρίσταστε. Θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις να θέσω για την πολιτική, την δασοκομική και τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σε σχέση με αυτή την πολιτική. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο στη συζήτηση για το αν ναι ή όχι πρέπει να ακολουθηθεί μία ή άλλη πολιτική. Χρειαζόμαστε όμως ανεξάρτητα αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία για την βιοπικιλότητα την δασική και κυρίως στοιχεία πληροφόρησης που θα βασίζονται σε κριτήρια αηφορίας και βιωσιμότητας. Χρειάζονται επίσης στοιχεία για τα δάση ως ε, ε, πηγές, ως ε, στοιχεία απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα. Χρειάζεται λοιπόν μια ανεξάρτητη επιστημονική βάση, ανεξάρτητη και αξιόπιστη, που θα καταφέρνει να είναι επαρκώ αξιόπιστη σε όλα τα κράτη-μέλη. Όταν κάνουμε λόγο για πιστοποίηση, δεν μπορούμε να αμελήσουμε ή να ξεχάσουμε ότι για πιστοποίηση απαιτείται ένα σύστημα ελέγχου, ελεγκτικό σύστημα επαρκώ ανεξάρτητο και αξιόπιστο. Θα ήθελα επίση να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Επίτροπο Ποια είναι η τοποθέτηση, ποιο ποσοστό σε σχέση με τη δασοκάλυψη ε, είναι εκείνο το οποίο ε, χρησιμοποιούμε. Είναι μια ιδέα αρκετά θα έλεγα που παρεκκλίνει πολύ. Εμείς στην Φινλανδία έχουμε 75% μια τέτοια δασοκάλυψη. Αν πρέπει ακόμα περισσότερο να πυκνώσουν τα δάση και να καλυφθούν και άλλες ε, εκτάσεις, τι θα γίνει με τους αυτοκινητοδρόμους, με τη στέγαση, με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και επιφάνειες. Θα πρέπει πολύ, πολύ συχνά να εγκαταλείψουμε λοιπόν τέτοιου είδους εκτάσεις ε, αν είναι να καλυφθούν με δάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και όντως πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις που θα έχουν οι αμερικανικές εκλογές. Ο νέος πρόεδρος είπε ότι θα αποσύρει τις Ηνωμένες από τη Συμφωνία του Παρισιού. Επίτροπε. Για την αναδάσωση. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, στη Ρουμανία Φερρυπίν, ε, υπάρχουν προβλήματα νομοθετικής φύσεως. Παρότι υπάρχουν κονδύλια για την αναδάσωση, Υπάρχουν οι δεσμεύσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διατήρηση των ε, δασικών εκτάσεων μέχρι το 2018. Δηλαδή, αν οι ιδιοκτήτε, α πούμε, θέλουν να δασώσουν δάση τα οποία είναι σε κακή κατάσταση, δεν μπορούν να το κάνουν. Σα παρακαλώ, μπορείτε να βρείτε μια λύση, ούτω ώστε να διευκολύνετε την αναδάσωση σε επίπεδο κρατών μελών που έχουν αναλάβει τι δεσμεύσει. Γιατί αλλιώ, ενώ έχουμε κονδύλια, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδάσωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσία σας, για την καταπολέμηση της αποψήλωσης των δασών και το σεβασμό των λειτουργιών των ευρωπαϊκών δασών. Χειροκροτώ τις καλές προθέσεις της δασικής στρατηγικής, καθώς και τα μέτρα που έχετε λάβει σε αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, επιτρέψτε να υπενθυμίσω ότι το κείμενο έλεγε στο πρώτο τμήμα τα εξής και παραθέτω. Η στρατηγική αφορά επίσης και το δασικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκειται στη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η βιομηχανία δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε επιμερισμένη αρμοδιότητα. Είναι ε, μια αρμοδιότητα για τη στήριξη που παρέχεται σε αυτήν την πολιτική δυνάμει του άρθρου 6 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται τώρα. Ε, με αυτό το θέμα ε, σε σχέση με, την, ε, με το δασικό κλάδο. Επίσης το κείμενο λέει πολλές φορές ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού, του δασικού κλάδου. Το ερώτημά μου λοιπόν το εξή. Πώς οι δασικές μας βιομηχανίες μπορούν να ανταγωνιστούν τις βιομηχανίες άλλων κρατών όπου οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ χάλια και όπου δεν υπάρχει κανένα σεβασμός του περιβάλλοντος πώ θα υπάρξει προστασία του περιβάλλοντο, ανταγωνιστικότητα και αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία και τα τρία. Επίση, διατήρηση των δασών είναι αξιέπαινη προσπάθεια. Αλλά ο κίνδυνο δεν είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράζεται και να υποκαθιστά τα κράτη-μέλη ε, στα διεθνή φόρουμ για τα θέματα των δασών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε πολύ καλά ότι 38% του γαλλικού εδάφους είναι δάσος. Και έχουμε 80 80.000 ε, συγγνώμη, εκτάρια το χρόνο, ε, όλο παραπάνω εκτάρια το χρόνο ε, αναδάσωσης. Ε, έχουμε 100.000 εργαζόμενους στον κλάδο κτλ. Εμείς έχουμε μεγάλες περιοχές ε, οικολογικές, ε, δάσο, οικολογικές τέτοιε περιφέρειε που είναι 80 στη Γαλλία. Αντί λοιπόν για την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα ήταν να στηρίξει τι εθνικέ στρατηγικέ για το δάσο. Δεδομένη τη ε, πολυπλοκότητα τη ευρωπαϊκή δασοκομεία, η κλιματική αλλαγή, η υποστήριξη του υπαίθρου, η πράσινη ενέργεια, η προστασία των δασών και των οικοσυστημάτων του, η βελτίωση τη ε, εκμετάλλευσή του είναι τεράστια διακυβεύματα για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα την κυριαρχία των κρατών μελών για ένα τόσο κρίσιμο τομέα. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγκίνες. Το συγγνώμη το Προεδρείο συνεδρίασε 6.30 γι' αυτό έφτασα καθυστερημένη. Ε, έχω δίπλα μου την ειδικό ε, ε, ε, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, Συναντήκατε με νέου γεωργού στην Ιρλανδία και συζητήσατε το θέμα τη διαθεσιμότητα γεών. Και σα είπαν ότι υπάρχει εξή σύγκρουση με την τάση οι να γίνονται δάση, να δασώνονται δηλαδή τι γίνεται το θέμα, το θέμα της χρήσης των δασών. Αποτελεί πλέον επίμαχο ζήτημα όχι μόνο ε, μεταξύ γενεών αλλά και, μεταξύ, αλλά και για γεωργούς οι οποίοι θέλουν περισσότερες γιες και δεν βρίσκουν με άλλους γεωργούς οι οποίοι ε, ασχολούνται με τα δάση, δασοκόμους δηλαδή. Ε, έχετε κάποια άποψη γι' αυτό, πώς μπορούμε να αυξήσουμε, να ικανοποιήσουμε αυτούς τους ε, ε νέους που θέλουν να γίνουν γεωργοί και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τα δάση. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο. Ε, πολλές οι ερωτήσεις. Τεράστιος ο αριθμός των σελίδων σημειώσεων του Επιτρόπου. Είναι αδύνατο πρόεδρε να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Δεν θα το προσπαθήσω θα αποσταλούν απαντήσεις ε, στους ευρωβουλευτές σε συγκεκριμένες ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα που διατυπώθηκαν. Όμως φυσικά η συνάντηση απόψε καταδεικνύει ότι υπάρχουν θέματα και αρμοδιοτήτων που τέθηκαν και σε σχέση με την παρέμβαση του κ. θέτει ένα ζήτημα το οποίο ε, υπερβαίνει θέματα πολιτικής όπως αναφέρθηκαν Έχουμε το θέμα της, των θέσεων απασχόλησης, το θέμα των ενεργειακών πολιτικών, των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα να πω στα μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση ότι ο Επίτροπος αναπτύσσει ένα ευρύτερο ε, έργο συντονισμού πολιτικών για αυτά τα θέματα. Θα ακουστούν λοιπόν για αυτά τα θέματα οι παρεμβάσεις ειδικέ του σε σχέση με το πώς ε, ε, το ενεργειακό μείγμα και άλλα συναφή θέματα έχουν ε, επιπτώσεις. Θα υπάρχει ευκαιρία λοιπόν να δούμε την ε, πολιτική προοπτική, πώς εντάσσεται η δασοκομική πολιτική στις διάφορες πολιτικές της Ένωσης. Θέλω σε σχέση με την κυρία Κρέστιγκερ, η να την ευχαριστήσω για τις προσπάθειές της. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχουν θέματα που οδηγούν σε κάποιες συμφωνίες, υπάρχουν όμως και διαφορές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την αναδάσωση δυνατότητες υπολογισμών, ποσοστού δασοκάλυψης όπως αναφέρθηκε και σε σχέση με την Φιλανδία και σε σχέση και με άλλες χώρες που βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση και έχουν αντίστοιχα μελήματα και ανησυχίες και για τον δασοκομικό τομέα και για την LULUCF και για τις ε, ε, δυνατότητες διαχείρισης ε, της δασοκομείας. Όλα αυτά είναι θέματα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δια, διαμορφώνει προτάσεις ε, είναι θέμα αξιολόγησης ε, και να δει κανείς πώς στον δασοκομικό τομέα μπορεί με 73% δασοκάλυψης π.χ. στη Φινλανδία και δασοκομικών δραστηριοτήτων να δει κανείς το διαφορετικό τοπίο που υφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι δεν υπάρχουν αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη, πάρα πολλά κονδύλια δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ε, πτυχές αυτές και για τη δημιουργία απασχόλησης. Είναι λοιπόν θέμα να δούμε πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια σε σχέση για παράδειγμα με την ανάπτυξη της υπαίθρου και πρέπει να δούμε ότι εφόσον ε, σε σχέση με την ε, νομοθεσία μπορεί κάποιες πτυχές να μην καλύπτονται πρέπει να δούμε τι μπορεί όμως να γίνει για να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Υπάρχει σημαντική συνεισφορά για το μείγμα πολιτικών που μπορεί να συνεισφέρει για την ε, αηφορία. Όσον αφορά για τα θέματα της ε, ε, τα θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Δασοκομείας που υποστηρίζει αυτό το έργο και που στις δράσεις ε, που έχουν αναλυφθεί στη μόνιμη επιτροπή για παράδειγμα εξέτασης των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων θα υπάρξει μια αναθεώρηση, ενδιάμεση αναθεώρηση των πολιτικών αυτών για τη δασοκομεία και θα υπάρξει έτσι μια ευκαιρία να ξαναδούμε και να αναθεωρήσουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα και τι πρέπει να γίνει οι κανονισμοί σε σχέση και οι διατάξεις ε, ε, με την Ρουλουσίεφα και την επικαιροποίησή τους η πρόταση αυτή επικεντρώνεται στις ε, εκπομπές ρήπων που είναι ανθρωπογενείς ε, και πρέπει να δούμε κατά πόσον λοιπόν μπορούν να αναλυθούν ε, δράσεις για την βελτίωση της κατάστασης ακολουθούν τις ε, κατευθυντήριες γραμμές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου και σε σχέση ε, με τον ε, συνομοθέτη αυτόν και σε σχέση με τις διαφορετικές απόψεις που υφίστανται θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν και αρκετά άλλα θέματα σε σχέση με τον κύριο Φράνεγκαν που ανέφερε για παράδειγμα την το θέμα των ε, δασών σε σχέση με ε, περιοχές που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ε, απομόνωσης της υπαίθρου. Και πρέπει όλα αυτά τα θέματα να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να ληφθούν υπόψη σε σχέση με δράσεις μέτρα αναδάσωσης για παράδειγμα που πρέπει να αποτελούν και αυτά ένα μέρος της δράσης μας να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι φυσικά μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν από πλευράς νομοθετικών πρωτοβουλειών, όπως για παράδειγμα για τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Το 7ο πρόγραμμα δράσης από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σφαιρικά και για την Ινδονησία που ε, τέθηκαν κάποια ερωτήματα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την αηφορία για προϊόντα τα οποία ε, παράγονται μετά από την αποψήλωση δασών στην Ινδονησία, Μαλαισία και σε άλλες ε, χώρες του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σε σχέση με, αυτές, με αυτά τα θέματα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ελευθέρου εμπορίου διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο ώστε να μπορούν να υλοποιούνται οι διατάξεις αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και για τη χρηματοδότηση για παράδειγμα για τη συνδρομή που μπορεί να παρασχεθεί στην ε, Ινδονησία για την πιστοποίηση της ξυλίας που εξάγεται από αυτή τη χώρα λαμβάνοντας υπόψη τον, ε, την πτυχή της αηφορίας ε, σε σχέση με οποιαδήποτε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ε, για την Ινδονησία αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι ζωτικό θέμα. 4 δις ε, ευρώ εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένδειξη του μοχλευτικού αποτελέσματος που μπορεί να επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δράσεις της. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό και θέλουμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα με τη δράση και την πολιτική μας. Η νέα πολιτική για την, ε, βιο, την βιομάζα και την ε, βιοενέργεια ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζει και τα μελήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών και για την βιοδιαχειρισιμότητα και βιωσιμότητα σε σχέση με τη δράση διαφορετικών γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τη συνιστόσα αυτών των πολιτικών σε σχέση με τη βιοενέργεια και τη βιομάζα όσον αφορά την ε, εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί σε σχέση με τους πόρους. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα που πρέπει να μπορέσουν να ολοκληρωθούν, να μπορέσουν να ολοκληρωθούν κατά το άμεσο μέλλον και όσον αφορά το cascading, την κλιμακούμενη δράση και επιπτώσεις, ε, η πολιτική αυτή σε σχέση με την χρήση των ε, δυνάμεων της αγοράς ε, μπορεί να καταδείξει ότι υπάρχει ένα ζήτημα και προβλήματα που δημιουργούνται όσον αφορά τη διασπάθηση των φυσικών πόρων, για παράδειγμα της ξυλίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα ειφορίας. Εξετάζουμε αυτά τα θέματα σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις τους και θα παράσχουμε προσανατολισμούς όσον αφορά την, ε, τις δραστηριότητες αυτές ε, και τις ε, δικές μας δράσεις και στην ε, Γενική Διεύθυνση από πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την βέλτιστη χρήση της ξυλίας. Εδώ υπάρχουν δυνατότητες ε, να συναγάγουμε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την βάση αυτή που έχουμε δεδομένων. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι κάλυψα σίγουρα γνωρίζω ότι δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις αλλά θα υπάρξουν απαντήσεις που θα αποσταλούν γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρεμβάσεις σας. Σίγουρα με τις σημειώσεις ε, που ε, λήφθησαν για την πολιτική που θα ακολουθηθεί, πρέπει να ακολουθηθεί, θα απαντήσουμε και θα τοποθετηθούμε από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επιτροπέ. Ο Επίτροπος και οι βοηθοί του σημείωσαν όλα σας τα σχόλια. Θα απαντήσουν γραπτός. Εγώ από την δική μου μεριά ε, και, από, και εκ μέρους του κύριου Μπούζεκ ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Μερικές φορές υποτιμούμε τα δάση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων και την κλιματική αλλαγή τουλάχιστον. Η διαχείριση των υδάτων είναι μία από τις ε, πιο σημαντικές ε, προκλήσεις του μέλλοντος. Επίσης, τα δασικά προϊόντα ε, χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, σε φάρμακα. Τα δάση επίσης αποτελούν χώρο κυνηγιού Τα κράτη-μέλη έχουν εθνικές πολιτικές, ανεπτυγμένες εθνικές πολιτικές. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη βιοπικιλότητα αλλά και μεγάλη ποικιλία εθνικών πολιτικών. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη τις ε, τοπικές συνθήκες. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει εθνικές πολιτικές, οπότε χαίρομαι που καταφέραμε και διοργανώσαμε αυτή την κοινή συνεδρία. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ την ε, γραμματεία και το προσωπικό μας για αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο κύριο Χόγκαν. Καλό βράδυ.